Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Καλή σας μέρα. Ο συνάδελφος Φιντσέντσο Ιόβινε με ενημέρωσε ότι εντάχθηκε στην ομάδα S&D. Τώρα, προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Καταρχήν, Έκθεση Winkler. Ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας.